Και έτσι τελείωσαν οι παρεμβάσεις του ενός λεπτού και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύντομη παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Αντζελίλη για την πρόληψη των ασθενειών που συνδέονται με την ηλικία στις γυναίκες. Η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, η έκθεση αυτή εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Έτος για, την, ε, ε, για ηλικιωμένα άτομα, για τη γύρανση του πληθυσμού, κατά ενεργό τρόπο που θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τα 27 κράτη-μέλη. Οι δημογραφικές εξελίξεις μας θέτουν ενώπιον πολλών προκλήσεων. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη ο, το ότι έχουμε 87 εκατομμύρια που υπερβαίνουν τα 65 έτη. Άρα η γύρανση θα μας απασχολήσει ε, ακόμα περισσότερο και ε, άνω των 80 έχουμε 1,3 και 1,6 εκατομμύρια αντιστοίχως άνδρες και γυναίκες. Παρά όμως το γεγονός ότι το προσδόκιμο ζωής για τις ε, γυναίκες είναι υψηλότερο από τους άνδρες πλήττονται από ασθένειες που επιδεινώνουν τη ζωή τους. Ιδιαίτερα όσον αφορά ε, καρδιακές παθήσεις καθώς και καρκίνο παθήσεις ε, του αναπνευστικού ε, κατάθλιψη και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και δυσκολίες πρόσβασης στις, ε, στα εθνικά σύστημα, συστήματα υγείας. Και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολλές φορές πρέπει να κλείνει κανείς ραντεβού και υπάρχουν ε, λίστες αναμονής που διαρκούν πολύ και αυτό αποθαρρύνει του ηλικιωμένου και ιδιαίτερα τι ηλικιωμένε. Μην ξεχνάμε ότι το 75,8% των γυναικών άνω των 65 ετών ζουν μόνες. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένε γυναίκες βρίσκονται στο κατόφλι της φτώχειας και βλέπουμε ότι το 24,5% των ε, γυναικών, των ηλικιωμένων γυναικών διατρέχει τον κίνδυνο φτώχειας. Και όπως ξέρουμε οι γυναίκες κερδίζουν κατά 17% λιγότερο από την αντίστοιχη ανδρική εργασία και πολλές φορές πρέπει να έχουν και μία παράλληλη δραστηριότητα για να συμφιλιώσουν την ε, οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική. Γι' αυτό το συνταξιοδοτικό καθεστώς είναι χαμηλότερο και δεν έχουν πόρους για μακροχρόνιες θεραπείες. Εάν λάβουμε υπόψη λοιπόν και τη γεωγραφική κατανομή θα πρέπει να προωθήσουμε το, τη, την καλή ποιότητα ζωής για τους ηλικιωμένους. Δηλαδή να υπάρχει μία σωστή υγειονομική περίθαλψη καθώς και πρόληψη έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι να, είναι, να ζουν μία καλή ζωή και να γίνεται και ο κατάλληλος προληπτικός έλεγχος. Από την πρόληψη λοιπόν μπορούμε να προωθήσουμε θέματα όπως την φυσική δραστηριότητα, ε, την καταπολέμηση της χρήσης αλκοόλ και καπνού και σύμφωνα με τον ΠΟΗ, οι γυναίκες που καπνίζουν θα ανέλθουν από 12 σε 25% το 2025. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο για να μην υπάρχει κοινωνικός ε, αποκλισμός που δημιουργεί και ενισχύει την κατάθλιψη. Ευχαριστώ κύριε Αντζελίλη. Περνάμε σε δικασία και HDI, οπότε έχουμε πέντε συναδέλφους που επίλυσαν ενδιαφέρον. Ακούμε πρώτα τον κύριο Λουχάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, η σκλήρινση κατά πλάκας πλήττει κυρίως τις γυναίκες. Πρόκειται για μία νευροεκφυλιστική νόσο η οποία πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες άνω των 65 ετών. Ε, Ζητήσαμε λοιπόν να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και η Κομισιόν θα πρέπει να προωθήσει την ίση πρόσβαση των γυναικών ε, σε υγειονομική περίθαλψη όταν μιλάμε για ασθενείς με σκλήρινση κατά, πλάκα, Θα πρέπει λοιπόν να Υπάρχει ιδιαίτερο εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό σε κάθε χώρα για να αντιμετωπιστεί σωστά αυτή η ασθένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσικά. Ευχαριστώ. Μέσα στα πλαίσια της αντιμετώπισης των ηλικιωμένων και της συμμετοχής στην ενεργό ζωή θα πρέπει να υπάρχει μία ενσυνειδητότητα των ε, προβλημάτων που σχετίζονται με την προχωρημένη ηλικία. Δυστυχώς οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο ε, από μακροχρόνιες ασθένες. Το 75% των γυναικών κάθε, πάνω από 65 ζουν μόνες και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ Υπάρχει και το πρόβλημα των αγροτικών περιοχών όπου η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι περιορισμένη. Δεν υπάρχουν νοσοκομεία που να δέχονται επίγοντα περιστατικά. Γι' αυτό χρειάζεται, ε, χρειάζεται περισσότερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές. Σας ευχαριστώ κυρία Βέτμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρώπη λόγω της ε, αυξανόμενης, ε, του αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής ε, φαίνεται πως έχει ένα πληθυσμό ο οποίος γυράσκει ειδικά και σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπάρχουν επίσης γυναίκες οι οποίες ζουν κατά πολύ περισσότερο από, τις, ε, από τους ε, άντρες και πάνω από 50 εκατομμύρια από αυτές είναι πάνω από 76 ετών. Λογικό είναι λοιπόν πως πρέπει να αναπτύξουμε τις ανάλογες στρατηγικές επικοινωνίες γιατί το να γυράσχει κανείς χωρίς ε, δραστηριότητα δεν κοστίζει μόνο την υγεία του ίδιου του άντρα ή της γυναίκας αλλά κοστίζει σε ολόκληρη την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία Γιαζαβέσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε όλοι πως οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες, αλλά δεν γνωρίζουν όλοι πως μετά την ε, σύνταξη οι γυναίκες ε, έχουν χειρότερη υγεία και μετά από τα 65 οι γυναίκες ε, είναι πιο ευάλωτες ε, στις ε, αρρώστιες του γύρατος, ειδικά τώρα όπου οι κυβερνήσεις ανεβάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης χωρίς να σκέφτονται το τι θα γίνει με τους ε, ηλικιωμένους. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμάσουν τον κόσμο για την γύρανση. Η πρόληψη μπορεί να βελτιώσει και τη σωματική και την πνευματική υγεία και αυτό θα πρέπει να αισθηθεί ιδιαίτερα στις γυναίκες γιατί έχουν διπλό πρόβλημα και υφίστανται διπλές διακρίσεις και από την οικονομία γιατί πληρώνονται λιγότερο αλλά και επειδή ασθενούν περισσότερο στην τρίτη ηλικία. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ και την κυρία Αντζελίλη για την έκθεσή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η υγεία είναι σημαντική κυρίως για τις γυναίκες οι οποίες ζουν περισσότερο από τους άνδρες. Έχουμε λοιπόν καθήκον να εξασφαλίσουμε την καλή κατάσταση υγείας των γυναικών μέσα από καλές ε, θεραπευτικές μεθόδους έγκαιρη διάγνωση ώστε να αξιοποιήσουν οι γυναίκες όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρονται. Οι προληπτικές εξετάσεις είναι διαθέσιμες σε, στις περισσότερες χώρες αλλά οι πολλές γυναίκες δεν τις εφαρμόζουν και αυτό ισχύει κυρίως για τις μαστογραφίες. Δεν χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που υπάρχουν και αυτό είναι θλιβερό διότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί πάρα πολλές ε, καταστάσεις. Ευχαριστώ κυρία Σάρη. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ το θέμα της υγείας ε, των ε, ηλικιωμένων είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί, ειδικά σε μια κοινωνία η οποία γυράσκει. Η ζωή μας βεβαίως επιμικίνεται, αλλά πρέπει να υπάρξει και πρόληψη των ασθενειών, η οποία δυσκολεύει λόγω της ε, οικονομικής κατάστασης. Το επίπεδο των συντάξεων και εισοδημάτων των γυναικών είναι συχνά πάρα πολύ χαμηλό, οπότε δεν έχουν ιατρική κάλυψη συχνά. Επιπλέον, οι γυναίκες συχνά ε, φτάνουν σε ένα σημείο να ζουν μόνες τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουν υπόψη και να συζητηθεί δημοσίως. Το ζήτημα λοιπόν της ε, γύρανσης των ε, γυναικών και τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που προκαλεί. Δεν βλέπω λοιπόν, να ζητάει κάποιος άλλος τον λόγο στην διαδικασία και της ΔΙΑΗ. Οπότε θα δώσω τον λόγο στον κύριο Επίτροπο για να τοποθετηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Επίτροπο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λίγα λόγια στα Ιταλικά στην κυρία Αντελίνη. Την ευχαριστώ για την έκθεση αυτή, την εκτενή αυτή έκθεση, η οποία θα συνεισφέρει στις ε, προσπάθειές μας να βελτιώσουμε την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και ιδιαίτερα των γυναικών. Και καταρχήν θα πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι πολλές από τις ανησυχίες που εκφράζονται, που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση και εκεί που μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο θα πρέπει να το κάνουμε. Και τώρα θα περάσω στα αγγλικά. Η έκθεση, κύριε Πρόεδρε, δείχνει σαφώς ότι υπάρχουν ασθένειες που προσβάλλουν τις γυναίκες, κυρίως όπως η οστεοπόρωση που επικρατούν, ασθένειες που επικρατούν μεταξύ των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ και αυξάνονται και ορισμένες παθήσεις όπως οι καρδιαγγειακές και ο καρκίνος του πνεύμονα. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Το φύλλο είναι παράγοντας ισότητας και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις πολιτικές μας για την υγεία. Επιτροπή ε, ασχολείται σοβαρά με αυτό το θέμα της χρόνιας παθήσεις ε, και την γύρανση του πληθυσμού στις κοινωνίες μας που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα της υγείας διότι όπως όλοι είπαν στις παρεμβάσεις τους οι Ευρωπαίοι ζουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 25% της ε, ζωής μιας γυναίκας ωστόσο διανύεται κάτω από συνθήκες κακής υγείας. Υπάρχουν δε επίσης και οι χρόνιες παθήσεις που δύσκολα αντιμετωπίζονται, γι' αυτό πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι χρόνιες παθήσεις είναι αναπόφευκτη συνέπεια της διαδικασίας της γύρανσης. Πάρα πολλά μπορούν να γίνουν για να προλάβουμε ή να, μετριάσουμε αυτές τις χρόνιες παθήσεις. Όλες δεν είναι δυνατόν να προληφθούν βεβαίως, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν κάνουν πολλά πράγματα για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να κάνουν υγιείς επιλογές για τον τρόπο ζωής τους. Και η στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2010-2015 περιλαμβάνει την υποχρέωση να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς τα θέματα υγείας μέσα από τις κατάλληλες πολιτικές κάτι με το οποίο ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η στρατηγική πρέπει να προωθεί, να προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση για την ισότητα στον τομέα της υγείας, με έμφαση στο κάπνισμα, το ε, ε, AIDS και τον καρκίνο. Και γίνονται προσπάθειες για ε, συνεργασία μέσα από κοινέ προσπάθειες και κοινού πόρους. Εφαρμόζονται σχέδια δράσης ήδη με, που εστιάζονται σε καινοτόμους ε, λύσεις όπως το Care and Cure, να προλάβουμε και να θεραπεύσουμε και έχουν γίνει και πάρα πολλές άλλες δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες. Η Επιτροπή ε, εστιάζεται στην πρόληψη των ασθενειών σε πολλούς τομείς μέσα από διάφορες προσεγγίσεις. Η πλατφόρμα για την διατροφή, τη δίαιτα, τη σωματική δραστηριότητα, οι εργασίες για την υπερβολική κατανάλωση υνοπνεύματος ε, και οι προσπάθειες για την ε, διακοπή, για την εγκατάλειψη του καπνίσματος. Ε, υπάρχουν δυστυχώς σε πάρα πολλές χώρες όλο και περισσότερο γυναίκες που καπνίζουν, νέες γυναίκες κυρίως και οι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία αλλάζουν και πρέπει λοιπόν να προσαρμόζουμε αντίστοιχα τις πολιτικές και τις δράσεις μας θα αρχίσουμε σύντομα να δουλεύουμε πάνω σε ένα πρόγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη τη διάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη στους άνδρες και τις γυναίκες σε ό,τι αφορά τις καρδιαγγειακές παθήσεις και μια τελευταία παρατήρηση κύριε Πρόεδρε πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για τους προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο ε, του, ε, του, για τον καρκίνο του τράχυλου και των, ε, του εντερικού συστήματος. Έληξε η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση που είναι η έκθεση του κυρίου Αρία Ετσεβερία για την ε, ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς. Του δίνω το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ε, Καταρχήν